Συνόδου. Και επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 105, ο πρόεδρος της διάσκεψης των πρόεδρων των επιτροπών είπε ότι δεν υπάρχουν ενστάσεις στην Επιτροπή των Πρόεδρων των Επιτροπών όσον αφορά τις προτάσεις, συστάσεις της Επιτροπής ΕΚΟΝ για να μην υπάρξει ε, κάποια αντίρρηση σε κάποια εφαρμοστική και κατουσιώδηση πράξη. Αν δεν έχουμε ε, κάποια ένσταση μέσα σε 24 ώρες από κάποια πολιτική ομάδα, τότε θα θεωρηθεί ότι αυτές οι συστάσεις εγκρίνονται αλλιώς πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις συστάσεις